σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη αν καμιά φορά έτσι με συνεπέρνει η συζήτηση και παθιάζομαι. Συνήθως στο τέλος της συζήτησης γίνεται αυτό και όχι στην αρχή. Επιστρέφω στο κανονικό μου ύφος, στη φωνή και στον τόνο. Παρακαλώ, πρέπει να ε, εστιάσουμε στο Νότιο Σουδάν και σας ευχαριστώ που δεν χαλαρώνετε την προσοχή και διοργανώσατε αυτή τη συζήτηση. Ε, είναι ε, μια χώρα όπου οι ελπίδες τους έσβησαν μέσα σε λίγα χρόνια. Θα μπορούσε να είναι πλούσια, έχει πόρους φυσικούς. Αντίθετα, είναι πολύ δεινή η ανθρωπιστική κατάσταση. 30.000 αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να πεθάνουν από λοιμό και άλλες χιλιάδες που είναι ε, ε, σύμφωνα με το ΙΕ στα πρόθυρα του λιμού. Ε, ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι, πάνω από 700.000 έχουν φύγει από τη χώρα. Είναι από τις μεγαλύτερες προσφυγικές κρίσεις σήμερα και θα ήθελα να δούμε και τις άλλες προσφυγικές κρίσεις, όταν και αυτές συμβαίνουν εκτός των ιδίων μας συνόρων ή της περιφέρειας μας. Αθώοι πολίτες συνεχίζουν να υποφέρουν από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τουλάχιστον οκτώ τις τελευταίες, 80 τις τελευταίες εβδομάδες έχασαν τη ζωή τους και 150 από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου μαθαίνουμε. Και ε, μόνο στην πολιτεία Unity. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουν πρόσβαση. Η σεξουαλική βία κατά των γυναικών και των ανηλίκων έχει φτάσει σε συγκλονιστικά επίπεδα παρά τις δεσμεύσεις όλων των μερών στο Νότιο Σουδάν. Δεσμεύσεις για προστασία των πολιτών και για τερματισμό της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο λαός του Νοτιού Σουδάν δεν μπορεί να περιμένει. Η δικαιοσύνη και η συμφιλίωση θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών για να μπουν και τα θεμέλια για μια βιώσιμη ειρήνη. Για το λόγο αυτό καλωσορίζουμε την απόφαση της Αφρικανικής Ένωσης να ε, δημοσιεύσει το πόρισμα της Εξεταστικής ε, ε, Επιτροπής για να προχωρήσει στο δικαστήριο. Η νευτική Συμφωνία πρόσφατη είναι πραγματική ευκαιρία που δεν μπορεί να χαθεί. Είναι ευκαιρία για τον Νότιο Σουδάν να προχωρήσει προς μια διαφανή διακυβέρνηση υπόλογη που να θέτει το συμφέρον των πολιτών και του λαού υπεράνω όλων των υπολείπων. Και αν όλα αυτά εφαρμοστούν σωστά και η συμφωνία θα αποδώσει. Θα υπάρξουν μεταβατικοί θεσμοί για να μπορέσει να ανοικοδομηθεί η χώρα. Η κυβέρνηση έλαβε μια απόφαση να αυξηθεί ο αριθμός των ομοσπονδων πολιτιών, ε, αλλά αυτό αντιβαίνει και στο πνεύμα και στο γράμμα ε, της συμφωνίας. Το ίδιο ισχύει για την απροθυμία της αντιπολίτευσης να συμμορφωθεί με τα θέματα ασφαλείας. Ε, πρόσφατα στην πολιτεία Unity υπήρξαν ε, επεισόδια και είναι όλα πάρα πολύ ανισχυτικά γεγονότα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Ε, χτες στην Άντις Αμπέμπα έκαναν μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης οι πλευρές. Αυτό μας δίνει ελπίδες, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο τώρα το θετικό συμπέρασμα του διαλόγου και η θετική κατάληξη του διαλόγου ακόμα δεν διαφαίνεται. Μόνο η έγκαιρη εφαρμογή της συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική ειρήνη και τερματισμό των δεινών που υποφέρει ο λαός του Νοτιού Σουδάν για να σταματήσει και αυτή η ανθρωπιστική τραγωδία. Θα πρέπει ε, όσοι ε, αντιτίθενται σε αυτή την προσπάθεια από όλε τι πλευρέ να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παραμείνουν ατιμόρυτοι. Τώρα όμω τι πρέπει να γίνει, οπωσδήποτε και χειρία, επιγόντω. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, όλα τα εμπόδια να αρθούν για να υπάρξει πλήρης και ανεφόρον ανθρωπιστική πρόσβαση. Και υπάρχει μεγάλη ευθύνη για το κράτος, και τις κρατικές αρχές. Τώρα αρχίζει η δουλειά. Το South Sudan δεν μπορεί να Ανεχθεί να αποτύχει και αυτή η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Δεν το αντέχει η χώρα. Θα πρέπει να πιέσουμε για συνοχή καλωσορίζουμε τις ε, ε, συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης και της ε, επικοδομητικής τάσης των γειτονικών χωρών Σουδάν, Ουγγάντα, Αιθιοπία και Κένια. Ο Δόκτωρ Ζούμα και ο Αιθίωπας Πρωθυπουργός βοηθούν και εμείς έχουμε δεσμευτεί να βοηθήσουμε στην περιοχή αυτή η περιφερειακή ενότητα είναι εκ των όνων κάνευ. Υπάρχουν και άλλες προκλήσεις. Θυμίζω εχθές τα συμπεράσματα ε, ε, του σχεδίου δράσης για το κέρας της Αφρικής 2015-2020 και που ε, δείχνει ποια είναι η συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή εκεί. Χρειαζόμαστε επίσης και ένα ισχυρό όργανο που να παρακολουθεί η κοινωνία των πολιτών της χώρας με διεθνείς φορείς και περιφερειακούς. Υπάρχει μια κοινή ε, τέτοια επιτροπή. Ε, χαιρόμαστε για τον διορισμό του Προέδρου και πραγματικά θα ηγηθεί στην προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παραστέκεται στο πλευρό του λαού του Νοδίου Σουδάν κατά τη διάρκεια της μετάβασης από το Δεκέμβριο του 2013 που ξέσπασαν οι σειράξεις. Προσπαθούμε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να αρχίσει η πολιτική μετάβαση. Δώσαμε μαζική ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε πάνω από 116 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος η βοήθειά μας ήδη έχει φτάσει στα 107 εκατομμύρια ευρώ. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υπολογίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της μαζί με τα κράτη-μέλη έχουν χρηματοδοτήσει περίπου 41% του συνόλου της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Νότιο Σουδάν φέτος και μόνο και συνολικά 3,1 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι και ευάλωτοι ε, που τους δώσαμε βοήθεια για να σωθεί η ζωή τους ίδια. Αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ανθρωπιστική βοήθεια από μόνη της δεν αρκεί και δεν μπορεί να υποκαταστήσει ε, τους θεσμούς και την υγιή ε, διακυβέρνηση. Εμείς δεν δίνουμε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά υποστηρίζουμε και τους πέντε πυλώνες της συνευτικής βοήθειας από το Εθνικό Πρόγραμμα για το Αναπτυξιακό Ταμείο, αλλά για τους δύο πυλώνες διακυβέρνηση και ασφάλεια, η υποστήριξη θα έρθει από το μέσο σταθεροποίηση, σταθερότητα και ειρήνης και ε, την αφρικανική αντίστοιχη διευκόλυνση για την ειρήνη. Είμαστε τώρα έτοιμοι για να δουλέψουμε για μια μεταβατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, να ενισχυθούν οι θεσμοί και να ανοικοδομηθεί η χώρα σε γερά θεμέλια. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την ε, διαχείριση των ε, τεραστίων πόρων που διαθέτουν με ευθύνη και με δικαιοσύνη προς όφελος όλου του λαού. Η ε, Συμφωνία Κοτονού θα υπογραφεί για να επισημοποιηθεί η σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αυτό που επήγει είναι όλες οι πλευρές να δεσμευθούν ότι θα εφαρμόσουν τη συμφωνία. Αυτό είναι κομβικό, αυτό είναι κλειδί, το έχουμε συμφωνήσει με τις περιφερειακές δυνάμεις και είναι κοινό μας στόχος και κοινό ορίζον ε, στον προσανατολισμό μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω με χαρά να ακούσω τις απόψεις για τη συζήτηση αυτή που τη θεωρώ ε, τεράστια σημασία και πάρα πολύ χρήσιμα τα όσα εσείς συνεισφέρετε. Σας ευχαριστώ κυρία Ιπάτη. Και τώρα θα αρχίσει η συζήτηση. Πρώτος πρώτος ο κύριος Βέντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η σύραξη στο Νότιο Σουδάν είναι πολύ σημαντικό θέμα για την ομάδα μου. Η Νευτική Συμφωνία του Αυγούστου είχε θέσει ένα τέρμα στις εχθροπραξίες αλλά δεν έλυσε αυτό όλα τα προβλήματα της χώρας που αντιμετωπίζει τρομερή ανθρωπιστική κρίση. Ήταν απλώς το πρώτο σημαντικό βήμα προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Πρέπει να δεχτούμε με χαρά τις δηλώσεις των ηγετών του Νοτιού Σουδάν που δήλωσαν ότι θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι βιοπραγιών είναι πολύ σημαντικό αυτό με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε ως προς το ότι θα δοθούν αποζημιώσεις και σε παιδιά και για διοπραγές κατά γυναικών και παιδών. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα την πολύ σοβαρή ανθρωπιστική όπως είπα κατάσταση στη χώρα Δύο εκατομμύρια άνθρωποι χρειάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε υγειονομική περίθαλψη και οι αρρώστιες ε, είναι πάρα πολύ διαδεδομένες. Ελπίζουμε η αντίδραση της Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας να εμποδίσει, να βελτιώσει τα πράγματα εκεί, γιατί απειλείται και λοιμός. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λόγω της προσφυγικής κρίσης που ζούμε στην Ευρώπη αυτόν τον καιρό, έχει έρθει η ώρα τώρα της Συρίας και του Ιράκ. Αυτά κυριαρχούν στην επικαιρότητα, αλλά όπως είπε η Πατή Εκπρόσωπος, δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ότι υπάρχουν δύο κρίσεις εφάμιλες και σε διάρκεια και σε μέγεθος στην Αφρική, Κέντρο Αφρική, Γανική Δημοκρατία και Νότιο Σουδά. Μία χώρα με 30 χρόνια πολέμου που μόλις 4 χρόνια υπάρχει ως ανεξάρτητη και αυτή τη στιγμή έχει 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι ανθρωπιστικές κρίσεις που έχουν προκριθεί από τον άνθρωπο, είναι ανθρωπογενείς. Ο πόλεμος τα έχει φτιάξει αυτά. Και βασικά αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αφήσουμε πίσω μας τους πολέμους στο Νότιο ε, Σουδάν και να συνεισφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Αφρικανική Ένωση και περιφερειακές ε, ενότητες και με τη διεθνή κοινότητα έτσι ώστε να εδρεωθεί η Ειρνευτική Συμφωνία του Αυγούστου. Δεύτερον, θα πρέπει να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Μόλις το μισό των όσων ζήτησε ο ΙΕ εγκρίθηκε και δόθηκε από τους διάφορους δωρητές. Τρίτον, θα πρέπει με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε την επιστηστική κρίση. Και σύμφωνα με τη βαθμολογία του ΟΗΕ είμαστε σε κρίση επίπεδου 3, δηλαδή όλεθρος και καταστροφή. Δηλαδή θα πρέπει να εργαστούμε υπέρ της ειρήνης, υπέρ της χρηματοδότησης με περισσότερα χρήματα, να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική και επισητιστική κρίση και να υπάρχουν ε, διάδρομοι ανθρωπιστικοί για να φτάνει και η βοήθεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ από την ομάδα του. Κύριε Πρόεδρε, το 2011 το Νότιο Σουδάν έγινε ανεξάρτητο ε, και από τότε για πολύ κακούς λόγους ε, ε, ήταν πάντα στην επικαιρότητα. Χωρίστηκε λοιπόν σε δύο χώρες το Σουδάν και δυστυχώς λόγω της κατάστασης και της, των βιαιοτήτων μεταξύ των δύο τμήματων πολλά είναι τα εκατομμύρια των εκτοπισμένων και τα προβλήματα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμό είναι πάρα πολύ μεγάλα. Πριν από μερικέ μέρε ε, αναφέρθηκαν ε, κάποιε πρωτοβουλίε οι οποίε ε, είναι το αποτέλεσμα των προβολιών και των διαργασιών που είχαν ξεκινήσει το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι αλλά όχι υπερβολικά. Να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει η διαμεσολάβηση τη IGAD, αυτής τη κυβερνητικής αρχής, αλλά και της Αφρικανικής Ένωσης ε, γιατί από το Δεκέμβριο του 2013 ε, ο ντόπιο πληθυσμός ε, έχει υποφέρει πάρα πολύ. Δυστυχώς, δεν, δυστυχώς ο αρχηγός ο οποίος μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση δεν είναι πλέον μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Τρία λεπτά. Κύριος Τζέζεκ. Δεν είναι πολλά τα μέρη του κόσμου που αντιμετωπίζουν χειρότερες συνθήκες ε, από το Νότιο Σουδάν και όπου ο κόσμος ε, υποφέρει περισσότερο. Συμφωνώ ε, ότι, τον, ότι το κείμενο το οποίο υπεγράφει τον Αύγουστο είναι ένα θετικό κείμενο το οποίο ζητάει την επάυση του πυρός, ζητάει την, την απόδοση δικαιοσύνης, ε, κλπ. Ε, βεβαίως η δέσμευση των δύο πλευρών σε σχέση με αυτήν την συμφωνία δεν είναι αρκετά ισχυρή και η διαμάχη συνεχίζεται. Ο ντόπιο πληθυσμό είναι αυτός ο οποίος ε, υποφέρει περισσότερο εντό και εκτός των στρατοπέδων θα πρέπει να σταματήσει, να υπάρχει πάυση του πυρόσα, αλλά αυτό θα επιτευχθεί μονάχα εάν χρησιμοποιηθεί σειρά στοχευμένων δράσεων εναντίον της πολιτικής ηγεσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτεί το εμπάργκο των όπλων. Από την άλλη πλευρά και για να είμαι πιο θετικός, ε, η σημερινή έκθεση που δημοσιοποιήθηκε όσον αφορά ε, την έρευνα για το Νότιο Σουδάν, αυτό, Σουδάν, αυτό είναι όντως ε, κάτι θετικό. Ρωτώ λοιπόν κυρία Υπατή εκπρόσωπε, ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές του Νότιου Σουδάν θα ακολουθούν ακολουθήσουν την συμφωνία και με ποιο τρόπο θα λογοδοτήσουν οι υπέτη. Ε, αναφερθήκατε στην κοινωνία των πολιτών. Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί στενά με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών έτσι ώστε να καλύψει την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας ε, επιτόπου και ε, εάν ναι ποια είναι η στρατηγική. Από τώρα το λόγο έχει ο κύριος Χαβιέρ Κόουσο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, για άλλη μια φορά ε, συζητάμε για θηριωδίε. Πάνω από 50.000 είναι νεκροί, πάνω από 2 εκατομμύρια οι πρόσφυγε. και δεν είναι θεομηνία. Ε, η προϊστορία έχει σημασία. Δεν μπορώ ε, να ξεχάσω ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένε Πολιτείε πρόθεσαν την απόσχηση. Είναι περίεργο πώ δημιουργούν ένα δημιουργικό χάος ανάλογα όταν του συμφέρει. Εκεί είναι τα βασικά κοιτάσματα πετρελαίου για να μην μπορέσει να βάλει χέρι η Κίνα και να βαλκανοποιηθεί η περιοχή και ε, θυμάμαι και τα αντίστοιχα σχέδια. Αυτές οι θηριωδίες που έγιναν όθησαν ένα εμπάργο από τον ΟΗΕ ε, που εξακολουθούν ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε να το τηρούν ενώ κατά του Ισραήλ παραβιάζεται. Θα πρέπει ε, να ε, σταματήσουν οι μισθοφόροι και οι παραδόσεις όπλων, να ενισχυθεί ο περιφερειακός διάλογος, θα είπατε κι εσείς, και κυρίως να φροντίσουμε να μην βάλουν χέρι στα πετρέλαια που έχει εκεί, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ ξανά στον Πρασίνο. Ο κύριος ε, Ζόρντι Σεπαστιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πάτη εκπρόσωπε για την παρουσία σας. Σας βλέπω πολύ συχνά και αυτό σημαίνει ότι λαμβάνετε υπόψη και σας το αναγνωρίζουμε αυτό ευρύτατα. Υπήρξε μια συμφωνία ειρηνευτική που υπογράφηκε τον Αύγουστο, αλλά ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Συνεχίζουν ε, οι μάχες. 57 είναι νεκροί αρχές Οκτωβρίου, τα περισσότερα παιδιά. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας του Κοινοβουλίου και πραγματικά έχω τρομοκρατηθεί, έχω μείνει άναυδος από το που χρησιμοποιούν τις γυναίκες ως όπλο πολέμου. Γυναίκες και κορίτσια βιάζονται συστηματικά. Αυτό ω ε, ως Ευρώπη δεν μπορούμε να το ανεχόμαστε. Είμαστε ηθική ευτουργία αλλιώ. Χρειαζόμαστε να ε, διατηρηθεί ε, το εμπάργκο. Το Ισραήλ το παραβιάζει. όχι κυρώσει με ανθρωπιστική βοήθεια γιατί πλήττει το λαό αλλά πίεση για να υπάρξει αυτό το ανεξάρτητο δικαστήριο για να δικαστούν αυτοί οι άνθρωποι για εγκλήματα παγκόσμια ε, και να υπάρξει συμφιλίωση και αποζημίωση. Αν γίνουν όλα αυτά η Ευρώπη θα είναι παρούσα ε, και να ξέρετε κυρία Υπάτη εκπρόσωπε ότι είμαστε στο πλευρό σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ομάδας του το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κάρβερ. What's ο κύριος Κάρβερ δεν είναι εδώ. Micro, please. Okay. Italian translation. No Italian translation. Ναι, ήθελα απλώς ε, να πω ότι εδώ και πέντε λεπτά δεν ακούω την Ιταλική, ε, ε την, την Ιταλική διερμηνία. Δεν ξέρω, δεν, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ακροβατικά έτσι ώστε να προσπαθούμε να ακολουθήσουμε άλλη γλώσσα. Uh, Ωραία. Τώρα, εξ ονόματος ε, του FTD, ο κύριος Κάρβερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να έχει εμπιστοσύνη η Πάτη στο όργανο αυτό, διότι το 12 και το 2014 τα ελικόπτερα του ΙΕ είχαν στοχεύσει και ανθρωπιστικές πομπές. Αυτά δείχνουν κυρία Υπάτη μου ότι ο αντιπρόεδρος Ρικ Μακάρ ίσως δεν έχει τα μέσα της πολιτικής που δηλώνει. Τι δεσμεύσεις έχει αναλάβει η Ένωση ακριβώς για τον Νότιο Σουδάν. Υπάρχει καμιά εγγύηση ότι αυτά που λέμε μπορεί και να γίνουν. Ευχαριστώ. Thank you very much Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξ ονόματος της ομάδας CNF, το λόγο έχει ο κύριος Εντουάρ Φεράν.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 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατή Εκπρόσωπε. Είναι το πιο νεαρό έθνος ε, το Νότιο Σουδάν ε, και είναι μία από τις τελευταίες χώρες της Αφρικής. Μετά από δύο εκατομμύρια νεκρούς ε, και τέσσερα εκατομμύρια εκτοπισμένους, ενδεχομένως πνέει τα λίστια το Νότιο Σουδάν. Επομένως η βοήθεια είναι καλοδεχούμενη. Ωστόσο η χώρα αυτή θα πρέπει να γίνει βιώσιμη και βασίζομαι στις προσπάθειές σας για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε γιατί έγινε μεν συμφωνία ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνούμε την ιστορική βαρβαρότητα του ε, Χαρτούμ το οποίο δεν διστάζει να παρεμβαίνει ε, στρατιωτικά. Ε, Μη λησμονούμε επίσης ε, τον, το πλούσιο υπέδαφος και τον πλούτο σε πόρους αυτής της χώρας και θα πρέπει προσεκτική έτσι ώστε αυτοί οι πόροι να μην γίνουν τελικά η τελευταία σταγόνα ζωής για αυτή την περιοχή του κόσμου, για τον Νότιο Σουδάν. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μαρία Γκαμπριέλ. μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπατή εκπρόσωπε. Ναι, ε, επαγρύπνηση και διαρκής ε, ε, κινητοποίηση της, δημόσι... της διεθνούς κοινότητας. Τέσσερα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητη η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων και στα πλαίσια της συμφωνίας της 26ης Αυγούστου αλλά και το πρόσφατο υπογραφέν κείμενο της Αφρικανικής Ένωσης. δύο Ο ρόλος των περιφερειακών εταίρων ε, του Νοτιού Σουδάν αλλά και της διεθνούς ε, κοινότητας ε, θα πρέπει να παραμείνει σταθερός και η Αφρικανική Ένωση και η ΆΙΓΑΝΤ, η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη αλλά και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνεχίζουν <clears throat> να, να, συνεχίσουν να στηρίζουν τους εκτοπισμένους και αυτούς που απειλούνται από τον λοιμό. Τρίτο, ο αγώνας ε, κατά της ε, ατιμορρησίας. Ε, αυτό θα πρέπει να ισχύσει στην νότια, στο Νότιο Σουδάν αλλά και να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας στρατός ο οποίος θα είναι δημοκρατικός και σωστός έτσι ώστε να σταματήσουν αυτές οι σεξουαλικές και άλλες διαδικασίες παρανομίες τέταρτο Τώρα θα πρέπει να βοηθήσουμε την, τον Νότιο Σουδάν έτσι ώστε να ανασυγκροτηθεί και να επανικοδομηθεί με δημοκρατικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λίντα Μακάβαν. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπερτή εκπρόσωπε. Ε, ζητήσατε συγγνώμη τελειώνοντας, ολοκληρώνοντας την προηγούμενη συζήτηση γιατί μιλήσατε επαθιασμένα, μα όχι έτσι γίνονται σωστά τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν ε, σήμερα ε, θίγοντας το θέμα του Νότιου Σουδάν με πάθος να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια χώρα σωστή, να, να βοηθήσουμε τη χώρα να βγει από τις δυσκολίες. Αναφερθήκατε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, αναφερθήκατε σε χιλιάδες ε, ε, βιασμένες γυναίκες, σε χιλιάδες ε, νεκρούς αμάχους, σε εκατομμύρια εκτοπισμένους για, και άλλωστε μην λησμονούμε ότι η UNICEF και ο ΦΑΟ έχουν προειδοποιήσει για, για υπερχόμενο λοιμό ε, θα πρέπει οι συμφωνίες να γίνουν σεβαστές και κυρίως ε, να γίνει σεβαστή και να εφαρμοστεί η πάυση, ε, του πυρός. Πολλά μέτρα ακούστηκαν εδώ, εμπάργκο, όπλων κτλ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν κυρώσεις, όχι σε κυρώσεις οι οποίες να δημιουργήσουν πρόβλημα στον απλό κόσμο, κυρώσεις οι οποίες να αφορούν τους υψηλά ιστάμενους. Οι γυναίκες θα πρέπει να αποκτήσουν φωνή σε αυτή τη χώρα και πιστεύω πιστεύουμε ότι ε, τα μάλλα θα συμβάλλει αυτό στην ε, λύση της ε, κρίσης εάν, δεν, εάν παραμείνουμε απαθείς απέναντι στις εικόνες που βλέπουμε στην τηλεόραση, απέναντι στις γυναίκες που βιάζονται, τα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα για να βοηθήσουμε την Αφρική στο σύνολό της και τη χώρα αυτή ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φώτιγκα. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από μήνες αιματηρών σειράξεων, ο πρόεδρος τελικά υπέγραψε την Ειρηνευτική Συμφωνία που συνοδεύτηκε σε πολλές περιπτώσεις με παραβιάσεις του εκεχηρίας που είχε υπεγραφτεί. Είναι καλό να πιεστεί η χώρα από τους περιφερειακούς παράγοντες εκεί και από το Συμβούλιο Ασφαλείας καθώς και για την αποστολή μιας ειρηνευτικής επιχείρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά χρειάζεται συμφωνία στον ΟΗΕ για να εφαρμοστούν κυρώσεις διότι η δράση των αρχών του Νοτίου Σουδάν μας δείχνει ότι υπάρχει ακόμα πολύ κακοπιστία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την πειθαρχία σας. Σαφχάουζερ, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, 11 εκατομμύρια άνθρωποι εδώ αφορούνται. Αυτό είναι du chaos que του έμπολα. Εδώ υπό την ηγεσία των Αμερικανών δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Οι φυλές μεταξύ Αράβων και Ντίνκα συνεχίζουν τις διαμάχες. Υπάρχουν επίσης και θρησκευτικέ διαφορές μεταξύ των κατοίκων του Νοτιού Σουδάν. Πρέπει να διατηρηθεί επιτέλους η ενότητά του η αμερικανική πολιτική και η αφισβήτηση των συνόρων στηρίζεται και από την Ένωση με υποκρισία. Όλοι λένε, εγώ συνεχίζω να υποστηρίζω την ε, εθνική ενότητα. Μπορεί τελικά να γίνει και διέρεση της διαιρέσεως. Στην Αφρικανική Ένωση ξέρουμε αν μπορεί να βρεθεί μια λύση η μεταβατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας πρέπει να παραδεχτεί ότι η διέρεση του Σουδάν ήταν λάθος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βουλευτά. Ανδρέας Πλένκοβιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε. Μογκερίνη. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα ε, να καλωσορίσω την υπογραφή της συμφωνίας στη Τζούμπα μεταξύ των ε, κυβερνητικών ε, και των ε, ανταρτών. Με τον τρόπο αυτό θα σταματούσε, θα σταμάταγε αυτή η βία, οι πολιετήσε στην πιο νεαρά δημοκρατία της Αφρικής. Δυστυχώς όμως αδυναμητίστηκε αυτή η διαδικασία και έχουν ξαναρχίσει οι διαδικασίες ε, και έργα τα οποία, είναι, ε, τα οποία αντιτίθενται στην ε, συμφωνία. Οι δύο αντιτιθέμενες πλευρές εξακολουθούν να μάχονται. Επομένως, αυτό που θέλουμε είναι ενδυνάμωση των δημοκρατικών δυνάμεων. Επίσης, υπάρχει ανάγκη να βοηθηθεί ο πληθυσμός, αυτή η κοινωνία η οποία έχει υποφέρει κατά τη διάρκεια ε, της ε, σύραξης. Ε, είναι πολλά τα θύματα της βίας, είναι πολλές οι γυναίκες που έχουν βιαστεί, είναι πολλά τα παιδιά που έχουν απαχθεί. 300.000 ε, ε, συγγνώμη, είναι πολλά τα χρήματα τα οποία έχουν ε, δοθεί για την χώρα αυτή. Ωστόσο, 4 εκατομμύρια είναι οι άμαχοι οι οποίοι απειλούνται από την πείνα. Πρόκειται για μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στο Νότιο Σουδάν που πρέπει να λυθεί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άννα παρακαλώ. Η ανθρωπιστική κρίση στο νότιο Σουδάν, Σουδάν ε, είναι αποτέλεσμα ε, μιας ε, σύραξης η οποία έχει ξεκινήσει και έχει υποδαβλιστεί από περιφερειακούς ε, παράγοντες. Ε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και η διεθνής ε, κοινότητα δεν πρέπει να σιωπά απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση όπως έχει κάνει στο παρελθόν οι ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες στήριξαν ε, την ανεξαρτοποίηση του Νότιου Σουδάν το 2011 δεν είναι δυνατόν να αφιστούν και δεν πρέπει να αφιστούν προσπαθειών έτσι ώστε ε, να καταφέρουμε κάτι καλό ε, σε αυτήν την χώρα. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει άμεση πάυση πυρός στο Νότιο Σουδάν. Επίγει ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, είναι ε, πολύ οι ακροτηριασμένοι, είναι πολύ πολλές οι γυναίκες που έχουν βιαστεί, είναι πολλοί των οποίων απειλείται η ίδια η ζωή. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε στην χώρα αυτή να χρησιμοποιούνται γυναίκες και παιδιά σαν όπλα ε, πολεμικά. Ε, δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τη χώρα αυτή ε, να πυρποληθεί από άκρη σε άκρη. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει μπροστά σε αυτήν την βαρβαρότητα. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Ελπίζομαι, κυρία Μογκερίνη, η διαδικασία του χαρτούμ να οδηγηθεί εις πέρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα κύριος Μάρκ παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Νότιο Σουδάν είναι το πιο νεοσύστατο κράτος του κόσμου. Το 2011 όμως αυτό που ιδρύθηκε δεν ήταν κράτος. Ήταν μια βίαιη κλεπτοκρατία, εχμάλωτη στα νύχια τοπικών περιφερειακών συμφερόντων και συμμαχιών ε, διαφόρων ανταρτών και γητών κρατών. Μόνο τιμωρησία και φρίκη γνώρισε ε, ο πληθυσμό. Υπάρχει ενευτική συμφωνία και δεσμεύτηκαν τα μέρη να προχωρήσουν σε μεταβατική ε, διαδικασία. Αλλά εγώ έχω τι επιφυλάξει μου. Χωρί ισχυρή διεθνή παρουσία θα μείνει πάλι στα χαρτιά. Θα πρέπει ε, μαζί με του εταίρου μα να φροντίσουμε να σταματήσει αυτή η λαιλασία του πλούτου. Τα κλεμμένα θα πρέπει να επιστραφούν ή να παγώσουν γίνει ε, βιαιότητες, φρικαλαιότητες. Θα πρέπει να τιμωρηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πρωταγωνιστής και όχι business as usual. Αν χρειάζεται να επιβάλλουμε και κυρώσεις κατά των πρωταγωνιστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να είναι πάντα προσινής. Κατά τα άλλα, προσινής είναι μια λέξη που δεν συνήθισα ποτέ σε σχέση με το Σουδάν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος ε, Τζέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επατεκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για άλλη μια φορά έχουμε μια συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο για την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν. Πολλωστή, ποσοστή είναι, νιωστή. φλούμε. Τέλη Αυγούστου και πάλι είχαμε μια ενευτική συμφωνία μεταξύ των ηγετών των αντιπάλων στρατοπέδων Έχουμε από τη μια ε, το Ρίκ Μασάρ και από την άλλη τον ίν πρόεδρο Σάλβα Κύρ. Η ποσοστή συμφωνία ήταν από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος. Παρ' όλα αυτά, λέει, ότι εκπρόσωπο, συνεχίζονται οι θάνατοι. Αλλά είναι αυτός σκοπός πλέον εκεί η δολοφονία. Παιδιά σκοτώνουν. Δεν γνωρίζουν τίποτα παραπάνω τα παιδιά. Μια ολόκληρη γενιά έχει μεγαλώσει σε πόλεμο και βία. Και βλέπουμε ότι είναι πραγματικά ανθρωπιστική καταστροφή. Δεκάδες χιλιάδες λιμοκτονούν και από τη λειψιδρία και την ξηρασία. Υπόθηκε και προηγουμένως αυτό. Η τελευταία λοιπόν ενευτική συμφωνία μεταξύ των αντιμαχωμένων μερών προέκυψε μετά από ισχυρή πολιτική πίεση. Αλλά ο πρόεδρος Σαλβακή την ίδια μέρα που υπέγραψε ε, μίλησε για ε, επιβεβλημένη εκβιαστική συμφωνία. Δεν είναι καλό μήνυμα αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη και η Ένωση να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένε Πολιτείες και να επιβάλλουν κυρώσεις προς τους ηγέτες. Να μην το αποκλείουν. Εάν αυτή η νευτική συμφωνία δεν τηρηθεί, δεν εφαρμοστεί στην πράξη και δεν ε, δώσουν επιτέλους ειρήνη για τους πολίτες στη χώρα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η κυρία Κασέτου Κουέγγε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης για την πρόθεση της Συμφωνίας Ειρήνης στο Νότιο Σουδάν. Συμφωνία όμως η οποία απειλείται ε, από τις βιαιότητες ε, οι οποίες ε, συνεχίζουν στην νότια, στο Νότιο Σουδάν. Εκατομμύρια είναι οι Σουδανοί οι οποίοι υποφέρουν πλέον ενώ κινδυνεύουν και από ε, μεγάλη διατροφική ανασφάλεια η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε λοιμό. Η βοήθεια ε, είναι άμεση και απαραίτητη για τον ε, πληθυσμό. Κυρία Πρόεδρε, το Νότιο Σουδάν δημιουργήθηκε, γεννήθηκε μέσα από τα συντρίμια μιας, ενός εμφύλιου πολέμου αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό αυτό το κράτος να ζήσει χωρίς ειρήνη, διότι η ειρήνη δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς ε, την δικαιοσύνη. Επομένως, υβριδική, το υβριδικό δικαστήριο του Νότιου Σουδάν θα πρέπει οπωσδήποτε να επιληφθεί όλων των παραβιάσεων. Θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω την ε, κυρία Φερερίκα Μογκερίνη για τη θέση που έχει πάρει όσον αφορά την ειρήνευση στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μογκερίνη, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για το παθιασμένο και θετικό σας μήνυμα και τον επικοδομητικό σας ρόλο για την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν. Όπως, είπε, όπως είπατε και πριν, δεν πρέπει η κρίση των προσφύγων να μας αποτρέψει από το να βλέπουμε τι συμβαίνει αλλού όπως στο Νότιο Σουδάνο που πρόκειται για πραγματική τραγωδία. Πρέπει νομίζω να επιδειχθεί η κατάλληλη πολιτική θέληση ώστε να εφαρμοστεί η εκεχηρία. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευθεί και πρώτη μας προτεραιότητα να είναι η διασφάλιση μιας βιώσιμης και αξιόπιστης ειρήνης και η εφαρμογή της συμφωνίας του Χαρτούμ γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε κανέναν. Το Νότιο Σουδάν θα γνωρίσει τον λοιμό αλλιώς. Πρέπει να καταφέρουμε να επιστρέψουμε τη χώρα αυτή στην ειρήνη και την ασφάλεια και σε μια πραγματική εθνική συμφιλίωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ons. Μαριάς. Ο στρατός συνεχίζει να επιτίθεται στο Νότιο Σουδάν με καταστροφικά αποτελέσματα επί του πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει την αναπτυξιακή της βοήθεια για να καλύψει και το Νότιο Σουδάν έτσι ώστε να υπάρχει εγγύηση της ασφάλειας των περοσώπων η βοήθεια αυτή πρέπει δεν να φτάνει εκεί όπου πρέπει να φτάσει, όπου είναι οι περισσότερες οι ανάγκες. Δυστυχώς η σύραξη αυτή ήταν προβλέψιμη. Γιατί να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη παντού παγκοσμίω. Γιατί, γιατί οι προσπάθειες αυτές ειρήνευσης συστηματικά αποτυγχάνουν με τις αιματηρές συνέπειες που γνωρίζουμε δεν έχουμε πάρει μαθήματα φαίνεται. Ευχαριστούμε. Τελείωσαν οι παρεμβάσεις και τώρα θα αρχίσει το σύστημα της οφθαλμαθηρίας Catch ο κύριος Καπούτος. Ευχαριστώ πολύ. Επανειλημμένα συζητήσαμε ε, σε αυτήν την αίθουσα της Ολομέλειας, τη δύσκολη, μιλήσαμε για τη δύσκολη κατάσταση στο νότιο ε, Σουδάνα, όπου ε, η κυβέρνηση μέσω καταχρηστικών φυλακίσεων, πολιτικών ηγετών, μελών πολιτικών κομμάτων, δημοσιογράφων κλπ. ή μέσω βιαιοτήτων προσπαθεί να κάνει το δικό του νόμο. Το World Food το πρόγραμμα ε, αναφέρει ότι ε, τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα ενώ ε, εκατομμύρια είναι αυτοί που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν διατροφική ανασφάλεια. Πρόκειται για μια κυβέρνηση επίσης η οποία χρησιμοποιεί τα παιδιά και τις γυναίκες για να επιτύχει, σαν όπλα για να επιτύχει τους στόχους του. Σε κλίμακα από 1 έως 5 η κατάσταση κατάσταση ε, όσον αφορά την, το Σουδάν ε, για, την, ε, για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί είναι, έχει φτάσει ήδη στο 5. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Νότιο Σουδάν παρότι έχει πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές εν τούτης εκεί ο πληθυσμός του ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ταυτόχρονα από το 2013 βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των φυλών νουερ και ντίνκα. επιπλέον σύμφωνα με τον οηε το νότιο σουδάν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εκεί βρίσκεται σε κίνδυνο λιμού αυτή τη στιγμή υποσυτίζεται. επιπλέον 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός και εκτός της χώρας και έχουν πέσει μεγάλος αριθμός από αυτούς θύματα των νότιο σουδανών στρατιωτών. τη στιγμή λοιπόν που ο οηε κάνει έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή η ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να συμβάλλει στην οικοδόμηση του νέου νότιου σουδάν. παράλληλα θα πρέπει να υποστηρίξει τη δράση των ανθρωπιστικών οργανώσεων δίνοντας χρηματοδότηση για να παρέχουν τρόφιμα και υγειονομική περίθαλψη στον πληθυσμό. τέλος πρέπει να εφαρμοστεί η ειρηνευτική συμφωνία που υπογράφτηκε στην Αντίσαμπεβα αμπέμπα το μάιο του 2014 για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στα πολωνικά. Ε, κυρία Μογκερίνη, έχετε την πλήρη υποστήριξή μας στη δράση σας. Θα ήθελα όμως να σας καλέσω να στρέψετε την προσοχή σας σε δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι να ε, προσαχθούν στη δικαιοσύνη εγκληματίε. Εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια της Ευρώπης όπου πριν από 20 χρόνια περίπου ε, σοβούσε πόλεμο. και ξέρουμε τι εστί ατιμορρησία και ξέρουμε τι εστί δικαιοσύνη. Διότι εκείνοι ε, που βίασαν γυναίκες, παιδιά που έκαναν άλλα εγκλήματα πολέμου είναι εκείνοι που θα πρέπει οπωσδήποτε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Και κάτι άλλο που ήδη κάνουμε αλλά θα πρέπει να το ενισχύσουμε είναι το εξής συζητάμε να αρκούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να φτάνει σε όλους στο Νότιο Σουδάν όσοι πραγματικά το έχουν δεκρά ανάγκη. Ευχαριστώ ε, κύριε Γιάκοφσιτς. Και τώρα... Νικόλ Λεγκάς. Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν ε, ε, είναι ε, στην ουσία ε, η συνέχεια και ο αντίκτυπος ε, της απεικιοκρατίας. Η κατάσταση στο νότιο η Σουδάν εξηγείται από το πλούσιο υπέδαφος. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται αυτές οι μεγάλες αδελφοκτόνες σειράξεις οι οποίες κρύβονται πίσω από έναν δίθεν ε, εθνικιστικό ε, πόλεμο. Ξέρουμε ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται οι γίγαντες των πετρελαϊκών εταιριών. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν εταιρείε, συγκεκριμένη εταιρεία η οποία, έχει, η οποία εδρεύει στην Ελβετία και η οποία είναι εμπλεγμένη με πολλά φορολογικά και άλλα προβλήματα με απάτες πολύ μεγάλες. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει τουλάχιστον η προμήθεια όπλων στην χώρα αυτή, έτσι ώστε να σταματήσει ε, η κατάσταση. Ο κύριος Καστάλτο, παρακαλώ. Presidente, un raccolto annuale molto scarso, 30.000... 30.000 ε, είναι αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν να ε, πεθάνουν από την πείνα. Εκατομμύρια εκτοπισμένοι, εκατομμύρια σε διατροφική ανασφάλεια, ε, χιλιάδες, για τη, χιλιάδες γυναίκες βιασμένες, χιλιάδες παιδιά στρατιώτες. Εδώ δεν έχουμε ηγέτες που είναι καλοί ή κακοί, έχουμε αδίστακτους ανθρώπους ε, σε, χώρα, σε μια χώρα ε, η οποία δεν έμαθε τα διδάγματα του παρελθόντος με τις χιλιάδες νεκρούς ε, και τα εκατομμύρια <clears throat> εκτοπισμένους, τα θύματα δηλαδή του προηγούμενου πολέμου. Βλέπουμε έναν τεράστιο κατακαιρματισμό όσον αφορά το υπέδαφος, όσον αφορά την, τις εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να κερδίσουν από το πετρέλαιο της χώρας πολυεθνικές ιδιωτικές εταιρείες, ε, εταιρείες ε, οι οποίες στηρίζουν την ε, κατάσταση, εταιρείες οι οποίες προέρχονται και από την γυραιά Ευρώπη και που δεν θέλουν καθόλου να οδηγήσουν τη χώρα αυτή στα βήματα της δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε σε Άραβες, σε Κινέζους αλλά και σε Ευρωπαίους, σε εμάς τους ίδιους να συνεχίσουν αυτήν την κατάσταση. Εάν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα λάθη του παρελθόντος, τουλάχιστον να αποτρέψουμε τα λάθη του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε τη εκπρόσωπος κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη. Παρακαλώ. Θα, ε, δεν θα δείξω το ίδιο πάθος ε, σήμερα τώρα, όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει ε, αυτό το θέμα, αλλά γιατί πρέπει κανείς να δείχνει μια λογική, αλλά και γιατί Πραγματικά θεωρώ ότι η συζήτηση που είχαμε σήμερα το βράδυ εδώ είναι πολύ επικοδομητική ε, και μπορεί να ε, βοηθήσει. Από την ε, μία πλευρά είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με τον ρόλο που μπορούμε και πρέπει να παίξουμε. Ο ρόλος αυτός είναι στηρικτικός των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων και παικτών. Όλοι το αναφέρατε εσείς ότι είναι δηλαδή κάτι σημαντικό να συνεργαστούμε με τους τοπικούς, περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες. Ε, από πλευράς ε, ανθρωπιστικής ε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την εστίαση που έχουμε πάντα όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση και εμείς είμαστε μακράν ο πρώτος παρεμβαίνων όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση και όσον αφορά τους πρόσφυγες που μπορεί να προκύψουν από αυτή την κατάσταση ε, γιατί ανθρωπίνως ε, είμαστε κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνοι αλλά και γιατί μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλες αστάθειες στο μέλλον. Δεύτερον, όσον αφορά το πολιτικό σκέλος ε, και την ε, υλοποίηση της ειρήνης. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, εξαιρετικά ευαίσθητη και όπως είπα ε, και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση οι πολίτες του Νοτίου Σουδάν έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε αυτήν την συμφωνηθήσα ειρήνη οπωσδήποτε και από τις ε, δύο πλευρές και το είπατε και εσείς ε, υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν ε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέρον για τη μία ή την άλλη πλευρά. Θα πρέπει όλοι να αποδώσουμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες και ότι δεν θα υπάρξει ατιμορρησία. Ε, θα πρέπει κάποιος να πληρώσει οπωσδήποτε για, τον, για την οδύνη, για τον πόνο που έχουν ε, ε, περάσει οι πολίτες του Νότιου Σουδάν. Η κατάσταση είναι δύσκολη, γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τους τοπικούς παράγοντες Αφρικαρική Ένωση και την ΆΙΚΑΝΤ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία ε, Ήπατη εκπρόσωπε. Ε, σας λέγω λοιπόν